Μία ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς διαβίβασε την, ένα διορθωτικό κείμενο στο κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση το άρθρο 216, παράγραφος 4 του κανονισμού, αυτό το διορθωτικό θεωρείται εγκεκριμένο εκτός και αν μέσα σε 24 ώρες από την ακίνηση μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές ζητούν να ψηφιστεί. Το διορθωτικό υπάρχει στην ιστοσελίδα Seance en Direct και ο τίτλος θα δημοσιευθεί στα πρακτικά αυτής της Ολομέλειας. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη για την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Γκοτσολίνο. Θέτουμε σε ψηφοφορία την έκθεση, νέα ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες.